Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των παρεμβάσεων του ενός λεπτού. Συνεχίζεται αύριο η Ολομέλεια. Θα ξεκινήσουμε στις 9 το πρωί. Έχει ε, δημοσιοποιηθεί η μερίσια διάταξη. Είναι αναρτημένη στο σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρα στη συνεδρίαση.